Buenos días, Καλημέρα, λέει ο πρόεδρο. Σε όλε τι γλώσσε. Σιγά σιγά. Αγαπητοί συνάδελφοι, να προχωρήσουμε. Πρώτα τα σημαντικά. Έγκριση τη μερσία διατάξεω. Πάνω σε αυτό πρέπει να σας πω ότι το σημείο 4 όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση για τις ε, συνεχιζόμενες διαπραγματεύσει οργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις νομοθετικές διαδικασίες πρέπει να ζητηθεί μετά τις ψηφοφορίες, περίπου στις 11. Παρακάτω, το 10. Όσον αφορά την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων που είναι εισηγητής ο κ. Κοέλιο, αναβλήθηκε. Οπότε, η ψήφιση της ε, εκθέσεως Κοέλιο πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα, στο Στρασβούργο. 9 Δεκεμβρίου. Στις 18.45. Αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση, εγκρίνεται η ημερησία διάταξη και προχωρούμε στο δεύτερο σημείο ανακοινώσεις του Προέδρου. Πρώτα πρώτα. Σας υποβαλώ προς έγκριση την ακόλουθη σύσταση των συντονιστών. First, nomination of rapporteur, Mrs. Πρώτα απ' όλα θα ορίσουμε την εισηγήτρια που θα είναι η κυρία Γκόμες όσον αφορά ε, αυτήν την ε, σφαιρική γενική συνεργασία μεταξύ ενώσεις και των μελών από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά την Ινδονησία. Δεύτερον, η Μαρία Γαμπριέλ έχει οριστεί σύγκεντρια για δύο εκθέσεις σύναψη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά τη διευκόνηση για την έκδοση των διαβατηρίων και επίση για την συμφωνία μεταξύ Ένωση και Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά την επανεισδοχή. Καλώ. Οπότε εγκρίνονται οι συστάσει των ε, συνοριστών για αυτού του συζητά. και επίση να σα πω τώρα όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώ είναι βέβαια το γνωστό πρόβλημα του περιορισμού του χώρου και γι' αυτό και έχουμε ε, διερμηνία μόνο προς 12 γλώσσες. Συγγνώμη για όσους δεν θα έχουν ε, διερμηνία προς τη γλώσσα τους. At the room and thank you for your understanding. And we move on. Ευχαριστώ σας και τώρα προχωρούμε στην έγκριση των πρακτικών. Τα πρακτικά πρώτον της 3ης Οκτωβρίου και τις 17ης Οκτωβρίου ενεφόντος έτους. Εάν δεν έχετε κάποια αντίρρηση, εγκρίνονται τα προαναφερθέντα πρακτικά. Προχωρούμε τώρα στο πρώτο θέμα ουσίας. Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, πάρα πολύ κρίσιμο θέμα, μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, οπότε και θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδοτήσεως, το οποίο συνέταξε συνάδελφος κυρία Αντζελίδη. Έχεις προηγούμενη τροπή γυναικών και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι παρά την τεράστια σημασία του θέματος δεν υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιο νομοθέτημα ούτω ώστε να στηρίζει τα εθνικά μέτρα, τα εθνικά νομοθετικά μέτρα, ούτω ώστε να αντιμετωπίζεται η βία των γυναικών. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί σειρά ετών επιδιώκει το να υπάρξει κάποια νομοθεσία για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών. Αυτό ακριβώς και είναι το θέμα του σχεδίου γνωμοδότησης της κυρίας Αντζελίλη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παρουσιάσατε με πολύ μεγάλη ακρίβεια το πόσο κρίσιμη είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προφανώς γνωρίζουμε όλοι ότι η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις βασικές μορφές διακριτικής μεταχείρισης και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανέκαθεν λέγαμε σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο ότι πρέπει η βία να ε, υποβάλλεται σε ποινές. Ε, κυρώσεις μάλλον με, μέσα σε ποινικό πλαίσιο έτσι να καταπολεμηθεί με συγκεκριμένες ποινές αλλά επίσης έχουμε πει επανειλημμένως ότι χρειάζεται μια πολιτιστική επανάσταση στην οτροπία, στα ήθη και τα έθιμα, στις συνήθειες και στην ε, καθημερινή αντίληψη, διότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα πλήγμα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όχι μόνο σωματικής, αλλά και για την ισορροπία, την, τον αυτοκαθορισμό των γυναικών, τις οδηγεί στην απογοήτευση την ε, στέρηση της ελευθερίας και είναι ένας πραγματικός φραγμός στη συμμετοχή, την ελεύθερη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία. Από το 1999 ε, όρισε τη Διεθνή ημέρα για την ε, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ΟΗΕ, όμως το φαινόμενο δεν έχει την τάση να περιορίζεται. είναι γνωστά τα δεδομένα και δυστυχώς τα ποσοστά είναι σταθερά δεν έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια μεγάλες βελτιώσεις. Τα δεδομένα μας λένε ότι περίπου το 25% των γυναικών, δηλαδή μία γυναίκα στις τέσσερις στην Ευρώπη, έχει πέσει θύμα κακομεταχείρισης. Ε, μίας, ε, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της. Και τις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για σεξουαλική βία. Τώρα, ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο οργανισμό που είναι υπεύθυνο για το χάρτη αυτό εκπονεί μια έρευνα, μια πρόσφατη έρευνα για τη βία κατά των γυναικών. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε το Μάρτιο του 2014. Να σα πω κάποια στοιχεία εκ των προτέρων. Τι θα πρέπει να μα απασχολήσει. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία δείχνει ότι τέσσερις γυναίκες στις πέντε δεν ε, απευθύνονται σε κάποια υπηρεσία στήριξης ή βοήθειας μετά τη, αφού πέσουν θύμα ε, βίας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες που, πέσουν, ε, που θα πέσουν θύμα σοβαρότερης ή λιγότερο πράξης βίας θα απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές. Ή σε κοινωνικές υπηρεσίες ή σε κάποιον σε κάποιο φιλικό πρόσωπο. Πολλέ φορέ δεν μιλάνε με κανέναν. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο, Γιατί μα εξηγεί ότι το φαινόμενο τη βία κατά των γυναικών είναι κάτι που υποτιμάται. Είναι ένα φαινόμενο που αποσιωπάται. Πολλέ φορέ οι γυναίκε ούτε καν γνωρίζουν την νομοθεσία που ισχύει στο εσωτερικό ενό κράτου μέλου. Α μιλήσουμε για δύο γυναίκε στι πέντε. Περίπου οι μισέ από τι γυναίκε που πέφτουν θύματα κακομεταχείριση δεν γνωρίζουν σε ποιον απευθυνθούν. Δεν γνωρίζουν εάν το αδίκημα του οποίου έπεσαν θύματα ή η πράξη βία στην οποία επέστησαν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ε, ένα αδίκημα αξιόπινο. Αυτά είναι τα δεδομένα για το 2013 και μας εξηγούν πως και στην Ευρώπη είμαστε φρικτά καθυστερημένοι σε σχέση με την ε, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ιδιαίτερος ως προς την ε, οικογενειακή βία. Τώρα, συγκεκριμένες προτάσεις. Το Κοινοβούλιο ήδη έχει κάνει πολλά. Νομίζω ότι η θητεία αυτή κλείνει με ένα θετικό απολογισμό σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία και το Κοινοβούλιο θα μπορεί τουλάχιστον να πει ότι σε αυτή την πενταετία εγκρίναμε σημαντικότατες οδηγίες. Την οδηγία για τα δικαιώματα, τη βοήθεια και την προστασία των θυμάτων. Την οδηγία για την εντολή προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο την οδηγία για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και την προστασία θυμάτων, την ε, ε, οδηγία για την προστασία των ανηλίκων και την ε, παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο. Εδώ πρέπει να σταθούμε σε ένα νομοθετικό εργαλείο και αυτό να προετοιμάσουμε που να είναι αποδοτικό, αποτελεσματικό και προηγμένο ώστε να στοχεύσουμε συγκεκριμένα την βία κατά των γυναικών. Νομίζω ότι το κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να έχει τη φιλοδοξία να προτείνει μια οδηγία. Γνωρίζουμε ότι σε σχέση με τη νομική βάση έχουμε οπωσδήποτε και το άρθρο 84 σε ό,τι αφορά την πρόληψη της εγκληματικότητας, αλλά πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα. Πρέπει να στοχεύσουμε στην χρήση για την οδηγία που θέλουμε να προτείνουμε ε, να στοχεύσουμε στη χρήση του άρθρου 83 ως νομικής βάσης. Δηλαδή στόχος η βία κατά των γυναικών να συμπεριληφθεί μεταξύ των μορφών βίας που είναι ε, αξιόπινες και σοβαρότατες. Δηλαδή άρθρο 83. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί βεβαίως ομοφωνία από το Συμβούλιο. Ωστόσο, δεν είναι ένα στόχος που θα επιτευχθεί αυτομάτως, αλλά η βία κατά των γυναικών πρέπει να είναι προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο, γιατί είναι προτεραιότητα και για, προτεραιότητα και για τις Ευρωπαίες ε, πολίτες. Τις νέες ή και λιγότερο νέες γυναίκες της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει οπωσδήποτε να πετύχουμε το στόχο αυτό. Κλείνω λέγοντας ότι θα πρέπει στο μέγιστο βαθμό να αξιοποιήσουμε όλα τα νομικά εργαλεία που μας ε, διαθέτει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις επόμενες δύο προεδρίες, την ελληνική και την ιταλική, προκειμένου στο επίκεντρο της συζήτησης να τεθεί το θέμα αυτό. Να προσθέσω εδώ ότι κατά την άποψή μου ήταν σημαντικό να αποσπάσουμε τη συμμετοχή της Επιτροπής ΛΥΜΠ στην ε, προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Είμαστε η καθήλυνα αρμόδια, μάλλον η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή των Γυναικών, αλλά εδώ είναι πολύ καλό που συμμετέχουμε και εμείς γιατί χρειάζεται μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια. Το επαναλαμβάνω λοιπόν. Ο στόχος είναι ίσως δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά μπορούμε να τον πετύχουμε. Είναι στο παιδό μας και μπορούμε να φτάσουμε και να ζητήσουμε οδηγία. Ευχαριστώ. Relevant matter in which, in which is only, it is only obvious that despite national... προφανές πως παρά τις εθνικές στρατηγικές που έχουν κάποια κράτη-μέλη, Κάποια από αυτά είναι στην πρωτοπορία της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, αλλά δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί στην Επιτροπή μας. Προφανές λοιπόν και δικαιολογημένο ότι πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Αντζελίλη. Να συζητήσουμε. Η κυρία Χέτ, λοιπόν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα χιλιάδες γυναίκες στην Ευρώπη βιάζονται και υφίστανται βία γενικώ. Στηρώνονται ακόμα και εντός του γάμου κτλ. Και για να το καταπολεμήσουμε αυτό πρέπει να συνεργαστούμε και να εγκρίνουμε μέτρα στο τοπικό, στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αντζελίλη για το σχέδιο έκθεσης που εξετάζει το νομικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό επίσης το κείμενο για την επικουρικότητα και την αλογικότητα και τις εθνικές παραδόσεις να συμπεριληφθεί, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη να καταπολεμήσουν τη βία κατά των γυναικών. Δεν είναι δικαιολογία η επικουρικότητα για να μην κάνουν τίποτα. πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ μέτρων και προσπαθειών που αφορούν τις συνέπειες της βίας κατά των γυναικών και τα μέτρα που καταπολεμούν την ίδια τη βία. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τη βία κατά των γυναικών ή των ανδρών ως κάτι το οποίο είναι μια φυσική καταστροφή και δεν μπορεί να κάνει τίποτα η κοινωνία καταστροφή που πρέπει να δεχτούμε σήμερα. Περισσότεροι πόροι αφιερώνται στις συνέπειες της βίας αυτής. Περισσότεροι πόροι πάνε σε ανθρωπιστική βοήθεια και εκεί πέρα δεν επαρκούν, αλλά στην περίπτωση αυτή να για φυσικές καταστροφές. Ναι. πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση των γυναικών και να μιλήσουμε για τη βία. Όχι μόνο τις συνέπειες της βίας. Είκοσι κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση τη σχετική στην Επιτροπή της Κωνσταντινούπολης. Οπότε έχουν μέσα και νομοθεσία. Και το ερώτημα είναι το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνυπογράψει τη συνθήκη αυτή. Ένα άλλο ερώτημα και θα κατατεζώ. Και σχετική τροπολογία είναι τα παιδιά που βλέπουν αυτή τη βία που πρέπει επίσης να θεωρούνται θύματα του εγκλήματος. Και κάτι πρέπει να μπει και για τις ευπαθείς ομάδες. Ηλικιωμένοι μετανάστες ε, και τα εγκλήματα τιμής πρέπει να μπουν εδώ. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Σας ευχαριστούμε πολύ, ο Πρόεδρο. Υπάρχουν άλλε παρατηρήσει από άλλο συνάδελφο. Ο κύριος Ρομέρο. Η κυρία Ρομέρο. Πρόεδρε, όπως είπε και η προλαλή το πρόβλημα για κάποιο. είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Όχι μόνο θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση από πλευρά των κυβερνήσεων, αλλά επίση θα πρέπει να υπάρχει μια πρικοδότηση αντίστοιχη, ούτως ώστε να έχουμε κάποια ε, μέσα για να ληφθούν τα μέτρα για τις γυναίκες, οπότε θα πρέπει να θα γίνει με τα θύματα, γιατί ό,τι έχει γίνει δεν έχει μεταφερθεί στα κρατημέλη. Σε παραμένει το θέμα ταμπού σε πολλές χώρες, αυτό το θέμα της βίας, οπότε το ότι ακόμα δεν έχουμε κάποιο είδους ε, κοινή μεθοδολογία στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούμε να συνηθούμε για το τι, τι, τι προβλήματα μας απασχολούν, τι, τι, τι διαμετρήματος είναι. Αυτό είναι τεράστια δυσκολία. Και τελικά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ο ε, ορισμός καν του εγκλήματος. Τι θα πει βία κατά των γυναικών σε ε, κάποιες χώρες, δεν υπάρχει ο διαρκής χαρακτήρας, ας πούμε, παρά βέβαια το ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εγκρίνει ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα για τον ορισμό του εγκλήματος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δυσκολίες <coughs> όσον αφορά την περιχαράκωση που θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να βρούμε έναν ορισμό. Βεβαίως είναι και θέμα του να μαζέψουμε, να συλλέξουμε τα δεδομένα αλλά ε, αν μπορούσαμε θα έπρεπε να βάλουμε στη Eurostat μια τέτοια προτεραιότητα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάποια μεθοδολογία. Βέβαια τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλλά να μπορέσουμε να επιμείνουμε, να μαζέψει αυτά τα δεδομένα Eurostat να σταματήσει αυτό να είναι ταμπού. Ε, ε, έχουμε το, το παρατηρητήριο, το, το είπε και η Επίτροπος, αλλά τι έγινε, έγινε μια μελέτη. Ε, αυτό το είχαμε καταφέρει επί Ισπανικής Προεδρίας. Τι έγινε, ούτε ακούσαμε τίποτα. Ε, λίγο προχωρήσαμε. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την ουσία του προβλήματος. Και βέβαια ξέρουμε ότι πρέπει κάτι να γίνει, αλλά ούτε κοινή υπάρχει, ούτε πρόγραμμα δράση, ούτε ευρωπαϊκή στρατηγική. είναι αλήθεια ότι κάποια κρατημέλη θεωρούν το ζήτημα ταμπού. Οπότε βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της διαδρομής. Νομίζω θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να άρουμε αυτό το κενό που υπάρχει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο για να μπορέσουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Ευχαριστώ κύριε Ρομέρο και το έχει το λόγο κύριος Ευχαριστώ να συγχαρώ την κυρία Αντζελίλη για την εξαιρετική της δουλειά Συμμεριζόμαστε πλήρως το όραμά της και την ανάλυση της. Θα συμφωνήσω απολύτως με όσα ακούστηκαν ως τώρα. Απλώς ήθελα να σταθώ σε κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα. Ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει ίσως να επιμείνουμε περισσότερο είναι η δικαιολογία της νοοτροπίας, του πολιτιστικού παράγοντα. Η Ευρώπη έχει γίνει πολυπολιτισμική πλέον. Αυτό το θεωρώ πλούτο. Mm. Πρέπει αυτό να το ε, μετρήσουμε, να δούμε ότι είναι ένας παράγοντας θετικός και όχι κατερνητικό όπως κάποιοι πιστεύουν. Αυτή η πολιτιστική ανάμειξη, αυτό το αμάλγαμα είναι κάτι που μας προχωρεί. Από από την άλλη στις ευρωπαϊκές χώρες ακριβώς λόγω του πολιτισμικού στοιχείου η βία κατά των γυναικών πολλές φορές βρίσκει δικαιολογία σε θρησκευτικές ή πολιτιστικές αντιλήψεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει αυτό να το διορθώσουμε. Πρέπει το αδίκημα της βίας να οριστεί με σαφήνεια ώστε να αφορά όλους όσοι ζουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να έχουμε απουσία ορισμού που δικαιολογεί το αδικαιολόγητο. Συμφωνώ απολύτως με αυτό. Και δεύτερη παρατήρηση. Δεν ξέρω κυρία Ανζελίλη αν θα είναι ε, κάτι που μπορεί να καλύψει η έκθεσή σας, αλλά ίσως σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι να μπορούμε να πούμε και γι' αυτό. Οι χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας. Ιδιαίτερα των γυναικών στις χώρες εταίρους, σε πολλές χώρες εταίρους, και ακριβώς με πρόσχημα αυτό το πολιτιστικό ή θρησκευτικό στοιχείο, σε πολλές περιπτώσεις είναι φρικτή. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη ότι ακόμη και αν κάποιοι νόμοι έχουν ψηφιστεί σε κάποιες χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, λόγω χάρη για την κατάργηση της δουλείας, Ακόμη και σε χώρες όπως η Μαυριτανία ξέρουμε ότι η δουλεία συνεχίζεται. Όταν λοιπόν έχουμε απελεύθερους, δηλαδή ανθρώπους που απελευθερώθηκαν από το καθεστώς του σκλάβου, του βούλου, παρόλα αυτά το μυαλό τους παραμένει σε αυτό το νοητικό ε, πλαίσιο. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτό. Κυρία Αντζελίλη, λοιπόν, καλό θα ήταν να συνταχθεί μια τροπολογία για να αναφερθούμε και σε αυτές τις καταστάσεις. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσαμε... Σκέφτομαι ότι θα μπορούσαμε πολύ απλά να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό το, σε αυτό το τομέα. Θα μπορούσαμε στη Συμφωνία Συνδέσεις και Συνεργασίας, σε κάθε πρόγραμμα, να ζητάμε την ε, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το βρίσκω ενδιαφέρον. Και επίσης υπάρχει άλλη μια πτυχή. Δεν θέλω να είμαι προκλητικός, αλλά υπάρχει και το θέμα της γενετήσιας υγείας, της αναπαραγωγικής υγείας που βρίσκεται στο επίκεντρο όλης αυτής της συζήτησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι πολιτιστικές δικαιολογίες αρκούν. Και ήρθα, εδώ γιατί πιστεύω ότι δεν θα είμαστε αρκετοί άντρες στην αίθουσα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρωταρχικώς αφορά τους άντρες. Ήθελα λοιπόν να είμαι εδώ για να φανεί ότι και η δική μας μαρτυρία είναι σημαντική για το θέμα αυτό και ότι ενδιαφερόμαστε. Ευχαριστώ. Μένει, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάντοτε είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τον Λιμισελ. Έχει 100% δίκιο. Νομίζω ότι είναι θλιβερό το ότι δεν έχουμε τώρα περισσότερου για να το συζητήσουμε. Περισσότερου άντρε και περισσότεροι άντρε δεν τοποθετούνται πάνω σε αυτό, διότι ακριβώ όπω είπε και ο Λιμισελ αλλά και άλλοι, είπε με ένα μεγάλο τμήμα από αυτή την βία είναι και πνευματική, διανοητική, εκτό από σωματική, πολλέ φορέ συμπολιστική ή και θρησκευτική για φορά τι σχετικέ απόψει και Πάρα πολύ πρόσφατα ε, ε, είχαμε στον γάμο στη Μελβρετανία ε, τη γυναίκα σαν τμήμα της κινητής περιουσίας και εμείς επομένως που είμαστε τόσο πηγιοκρατική δύναμη Παρ' όλα αυτά είχαμε αυτή την άποψη ότι η γυναίκα αντικείμενο το οποίο υπόκειται σε καταπίεση, έλεγχο κλπ. Και πάρα πολύ πρόσφατα είχαμε μια πάρα πολύ προβεβλημένη ε, ε, υπόθεση που αποκαλύφθηκε δηλαδή ότι επί 30 χρόνια τρεις γυναίκες ε, ήταν φυλαγισμένες ως δούλες και γιατί αυτό παρουσίαζε τόσο ενδιαφέρον γιατί ήταν λευκέ. ενώ άλλε είναι φυλαγισμένες είναι σκλάβες, δούλες για λόγους θρησκευτικούς, για λόγους πολιστικούς αλλά κάνουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει, το αγνοούμε. Οπότε λέμε ότι για την πολυμορφία την γιορτάζουμε, την τιμούμε στην Ευρώπη και αυτό είναι η ισχύ μα και εντάξει όμως θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις προφάσεις ότι αυτό το λέει ο πολιτισμός μου, αυτό το επιβάλλει η θρησκεία μου, οπότε θα πρέπει επομένω να βρούμε τα χρήματα για να εντοπίσουμε το πρόβλημα, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι γίνεται και οι γυναίκες να έχουν κάποιες τηλεφωνικές γραμμές, κάποια, κάποια τηλέφωνα που μπορούν να καλέσουν και επομένω ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι θα πρέπει να βρούμε χρήματα, τέρμα πια τα λόγια και άρα κάτι να γίνει, κάτι να γίνει τώρα γιατί να σταματήσει ε, αυτού του είδους η ξαναγκαστική ε, διαδικασία του γενετήσιου ακροτηριασμού ε, αυτή η γάμοι που γίνονται κάτω των ηλικία 12, ξέρω ότι η κυρία Τζελίλη ε, έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά, έχει γίνει ε, την ομάδα υψηλού επίπεδου για, τη, για τις διακρίσεις επί τη βάση του φύλου. Όλα αυτά έχουν σχέση μεταξύ του, Πόσο μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχει σχέση και με την έκθεση τη πρωτοβουλία τη κυρία Λούνα, που θα συζητήσουμε αργότερα. Γιατί θέλουμε ακριβώ να μιλούμε για την προστασία των δικαιωμάτων, γιατί ή αυτό πανεπιευρώπηση δικαιωμάτων ή δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Are you willing to make another additional point, please? Ναι, θέλετε να πείτε κάτι άλλο, σύντομα παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Συμφωνώ με αυτό το οποία είπε ο άντρας συνάδελφός μας συμφωνώ. Πράγματι, εντάξει, υπάρχει θέμα με ανθρώπους που προέρχονται από άλλες χώρες και άλλες ε, θρησκείες, αλλά μην ξεχνάμε και την βία, την οικογενειακή. Δεν είναι μόνο σε φτωχά σπίτια, σε πλούσια σπίτια λευκών, σε κάθε χώρα στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να μιλάμε για τις χώρες αυτές του τρίτου κόσμου. Ας κοιτάξουμε πρώτα τι γίνεται μέσα στην Ένωσή μας. Κοιτάξτε, εγώ έχω ταξιδεύσει σε ολόκληρη τη Σουηδία και επισκέφθηκα διάφορα καταφύγια γυναικών. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται σε απλές καθημερινές οικογένειες και έχει αυξηθεί λόγω του κενού ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους. Ε, είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπατε, πολλές γυναίκες από τρίτες χώρες ε, ε πράγματι το υφίστανται αυτό, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τα του οίκου μας και πράγματι έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι άντρες σήμερα. Γιατί μπορούμε να το λύσουμε χωρίς άντρες. Of course, there have been women involved in this discussion. Πράγματι, και άντρες και γυναίκες συμμετείχαν στη συζήτηση γιατί αυτό είναι τραγωδία για ολόκληρη την κοινωνία στην οποία συμμετέχουμε όλοι. We just uh, mind the fact that although... Και βεβαίως ε, παρά το ότι τα κράτη-μέλη έχουν εθνικές στρατηγικές για τη βία κατά των γυναικών, επηρεάζεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δείχνει πως δεν διαφέρουμε πολύ, δεν διαφέρουμε όσο νομίζουμε, από διάφορες άλλες χώρες. Κάποιοι βλέπουν μόνο την καμπούρα των άλλων. Τα είπε ο κύριος Κάσμαν. Ε, σε πολλές χώρες η νόμιμη διακριτική μεταχείριση των γυναικών ήταν ε, ε πώς να πω, μέχρι χτες ας πούμε νόμιμο. Δηλαδή και η δολοφονία των ε, γυναικών ε, ήταν μια δολοφονία την οποία τιμωρούσε κανείς λιγότερο αυστηρά σε κάποιες χώρες. Κάποιες ε, χώρες έχουν ειδικά γραφεία της εισαγγελία, ε, της αστυνομίας, ειδικά για τα εγκλήματα κατά των γυναικών και χρειάζεται άρα ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία γι' αυτό και η έκθεση της κυρίας Αντζελίλη. Ε, θα σας δώσω το λόγο τώρα να συνοψίσετε πριν ε, περάσουμε στο επόμενο θέμα. στην διάταξη. Κύριε Αντζελίλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι συνοπτική. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Την συνάδελφο Χέντ, τον κύριο Ρομέρο, τον κύριο Κάσμαν, τον κύριο Λιμισελ. σας παρακαλώ να συνεισφέρετε με τροπολογίες, συγκεκριμένες τροπολογίες για να ενισχυθεί το κείμενο και να γίνει προφανώς πληρέστερο απλώς να υπογραμμίσω κάποιες σκέψεις. Η κυρία Ρομέρο θύμισε τη σημασία του να υπάρχουν επικαιροποιημένα δεδομένα, σαφή και συγκρίσιμα. Πρέπει να είναι προτεραιότητα της Eurostat αυτή. Χωρίς δεδομένα δεν μπορούμε να εργαστούμε σωστά, ούτε από νομοθετική σκοπιάς, ούτε από άποψη στήριξης κοινωνικών υπηρεσιών δεν μπορούμε να εργαστούμε όπως πρέπει, χωρίς δεδομένα. Επιτά συμφωνώ με την κυρία Χέντ ότι πράγματι τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, διατηρήσουν, να διαφυλάξουν την επικουρικότητά τους, όμως χρειάζεται οδηγία που να ε, ε, δημιουργεί μια κοινή πλατφόρμα. Αυτό θα ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για τις χώρες που από νομοθετικής πλευράς έχουν καθυστερήσει. Δεν έχουν όλες οι χώρες νομοθεσία ε, πρωτοπορίας, ούτε εντός ούτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκεφτείτε τη σύμβαση της Ισταμπούλ, της Κωνσταντινούπολης, επικυρώθηκε από τρία μόνον κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρία από τα 28. Άρα φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ Πρέπει να πω ότι ο νόμος πάντοτε χρησιμεύει. Να σας πω για παράδειγμα στη χώρα μου. Ο νόμος για την παρενόχληση, ένας καλός νόμος ε, πρωτοπορίας, δεν θα σταματήσει τον βίο άνθρωπο, το βίο άτομο που στο τέλος μπορεί να δολοφονήσει τη σύντροφό του, τη γυναίκα του, αυτόν που πραγματικά είναι είναι ζωώδης στη συμπεριφορά του και τον υποκινεί ένα ένστικτο βίας. Αλλά εντός εισαγωγικών όσοι σκέφτονταν να βασανίσουν τη γυναίκα τους, την πρώην γυναίκα, την πρώην σύντροφο, παίρνοντα συνεχώ γραπτά μηνύματα, περιμένοντα την κάτω από το σπίτι τη, ε, ουρλιάζοντα το τηλέφωνο. Αυτοί δεν το κάνουν πια. Διότι ξέρουν το βασανίσουν μια γυναίκα σέρνοντα 100 γραπτά μηνύματα την ημέρα, αυτό θα επιφέρει ποινικέ κυρώσει. Δεν το κάνουν πια, το κόψανε. Άρα πάντα ένας νόμος μπορεί να χρησιμεύσει. Ήταν λοιπόν ε, πολύ σωστά τα λόγια της κυρία Χέντ. Καλά και άγια όταν είπε ότι 25% των γυναικών ε, στην Ευρώπη έχουν υποστεί μορφή βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Αλλά εδώ δεν εννοούμε μόνον άτομα στο περιθώριο της κοινωνίας. Δεν μιλάμε για φτωχές μετανάστηδες που δεν έχουν άδεια παραμονής καν, για πρόσωπα που βρίσκονται σε δυσχερείς συνθήκες, ευάλωτες που είναι εκτεθειμένες. Και αυτές χρειάζονται φυσικά προσεκτικότατη παρακολούθηση, διότι εκεί που υπάρχει φτώχεια συχνά υπάρχει και περισσότερη βία, όμως είναι πάμπολες οι γυναίκες οι οποίες είναι επιχειρηματίες, ανεξάρτητες, πλούσιες και υποφέρουν, ε, πρέπει να υποστούν τέτοιες μορφές βίας. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις τείνουν να καταγγέλουν ακόμη λιγότερο αυτά τα φαινόμενα. Διότι κάποιος που δεν έχει τίποτα να χάσει πάει στην αστυνομία. Μια γυναίκα καριέρας φοβάται, φοβάται ξεκάθαρα ότι η αξιοπρέπειά της, η αξιοπιστία της μπορεί να μειωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αντζελίλη. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Επίσης ευαίσθητο, χάρτη πορεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη ομοφοβία και των διακρίσεων λόγω του γενετήσου προσανατολισμού και τη ταυτότητα του φύλου. Έκθεση τη συναδέλφου Λούνατσεκ. Σχέδιο έκθεση. «45 τροπολογίες έχουν υποβληθεί ω τώρα μεταξύ των οποίων κάποιε συμπληρωματικέ που προτάθηκαν από την ίδια την εισηγήτρια. Προτείνω να παραμένουμε σε δίλεπτες παρεμβάσει, αφού παρουσιάσει η εισηγήτρια το σχέδιο εκθεσή τη, διότι έχουμε ψηφοφορία στι στις 12.30. Με συγχωρείτε, στις 10.30. Στις 10.30. Και έχουμε ακόμη άλλο ένα σημείο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον χρόνο. Κυρία Λούνατσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μην ανησυχείτε. Ε? Από ό,τι πρόσεξα από την συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, υπάρχει φοβερός αριθμός, φοβερός βαθμός συνένεσης ως προς τις τροπολογίες. Δεν θα έλεγα ομοφωνία, αλλά μεγάλη τα ε, συνένεση. Ευχαριστώ λοιπόν τους τους εισηγητές για τη συνεργασία μας για το θέμα αυτό, καθώς και το προσωπικό της Επιτροπής, τη Γραμματεία. Ήδη την ε, πρώτη εξέταση την είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες, δεν θα ε, ανασταθώ λοιπόν σε όλες τις τροπολογίες, μην ανησυχείτε. Οι 23 από τις 45 τροπολογίες έχουν συνυπογραφεί από 5 πολιτικές ομάδες, εισηγητές 5 πολιτικών ομάδων. Για τις περισσότερες από τις υπόλοιπε, οι τέσσερις ομάδες τις συνυπέγραψαν, οπότε Μιλάμε για ευρεία συνένεση αυτή εξ αρχή και γνωρίζω ότι από το ΕΛΚ, του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ και την ΚΟΕ υπήρξαν κάποιε ανησυχίε για θέματα επικουρικότητα. Τι συμμερίζομαι τι ανησυχίε αυτέ και κάποιε όντω θα πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε προσεκτικά. Χθε είχαμε συνάντηση των σκιωδών και συζητήσαμε για το θέμα αυτό. Συμφωνήσαμε ότι από κοινού θα ε, υποβάλουμε συμβαστική τροπολογία την οποία αποστήλαμε χθε μετά τη συνάντηση των σκιωδών, την οποία θα ήθελα και να τη διαβάσω. Λέει 4α. Υπογραμμίζει ότι αυτή η συνολική πολιτική πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οργανισμών της και των κρατών μελών της ε, και των αρμοδιοτήτων που ορίζονται για αυτούς. Ε, με όσα άκουσα από τους σκιώδεις εισηγητές, ελπίζω ότι με αυτή τη συμβαστική τροπολογία θα είναι πολύ ξεκάθαρο τι, ε, πώς αντιμετωπίζουμε την επικουρικότητα και πώς αυτός ο χάρτης πορείας έρχεται να ενταχθεί σε κάθε επίπεδο λειτουργίας των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι λοιπόν ευχαριστήσω τους Σκιώδης και ίσως να σταθώ σε 4-5 τροπολογίες που υπευλήθησαν από άλλους συναδέλφους. Μία, η τροπολογία 5 του κυρίου Σκορία και του κυρίου Μπαρτολότσι, είναι η μόνη που δεν θα στηρίξω αυτή ως εισηγήτρια διότι πιστεύω ότι θα μπορούσε να ερμηνευτεί με τρόπους διαφορετικούς χωρίς να εντάσσεται στο συνολικό στη συνολική λογική της έκθεσης μια άλλη τροπολογία του κυρίου Οντί που εξηγεί τι θα πει LGBTI εντάξει αλλά μην φανταστείτε ότι όλοι το ξέρουν ότι είναι λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, ανθιφιλόφιλοι και διαφιλικοί Ε, έχουμε μια ε, τροπολογία για την ε, νέα στρατηγική που ζητάτε και του κ. Γιον, ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι ειδικοί περί και οι σχετικοί επαγγελματίε είναι εκπαιδευμένοι για θέματα LGBT. Είναι σημαντικό αυτό, <clears throat> γιατί και οι πρόσφυγες ξέρουν, πρέπει να ξέρουν τι ίσχυε για τις ε, περιπτώσεις LGBTI και στις χώρες τις οποίες φτάνουν. Για την ώρα αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ όλους. Ελπίζω στις 17 Δεκεμβρίου να έχουμε μια καλή πρώτη ψηφοφορία και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λούνατσεκ. Και τώρα η ώρα για τη συζήτηση. Κύριε Κάσμα, έχετε πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο γιατί φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία εδώ πέρα. συγχαρώ την Ουλρίκε για τη δουλειά που έκανε και να πω πως την στηρίζουμε. Επίσης θα ήθελα να επενέσω το έργο του ΕΛΚ που πραγματικά ασχολήθηκε με το ζήτημα και αναγνώρισε πως πρέπει να υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Υπάρχει οδικός χάρτης για τα πάντα εκτός από αυτό και αναρωτιέμαι γιατί ίσως μπορεί να εξηγηθεί η ντροπή του. Η ομάδα μου και εγώ έχουμε συνυπογράψει όλες και τις 41 Τροπολογίε για τι αρμοδιότητε που είπε η και Συμφωνούμε με την πρότασή της για μια συμβιβαστική τροπολογία. Δεν μπορώ να στηρίξω την τροπολογία 5. Ξέρω που, ποιο είναι το θέμα. Είναι το θέμα τη θρησκεία, αλλά υπονοεί πως υπάρχει μια ιεραρχία ε, δικαιωμάτων. Εντάξει, πρέπει να υπερασπιζόμαστε τη θρησκευτική ελευθερία, αλλά όχι το δικαίωμα να επιβάλλει κανείς την πίστη του σε άλλους, εάν έτσι μειώνονται δικαιώματα του άλλου. Και νομίζω πως εδώ πέρα υπονοούμε πως υπάρχει μία ανωτερότητα της θρησκευτικής πίστης. Ε, κοιτάξτε, η πίστη τα δικαιώματα είναι οριζόντια, όχι κάθετα. Κυρία Ματσόλα, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ουλρίκε για την παρουσίαση και τη συνεργασία που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως ξέρετε έχουμε συνυπογράψει τις περισσότερες τροπολογίες. Η έκθεση αυτή πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση και εκτιμώ τις προσπάθειες που έγιναν. Η ομάδα μας ε, θα το συζητήσει λεπτομερώς στις επόμενες ημέρες και αυτή τη στιγμή βεβαίως είμαι πολύ αισιόδοξη. Επίσης εκτιμώ το κείμενο που έχετε εδώ πέρα για την επικουρικότητα. Οπότε συμπερασματικά ελπίζω να συνεχίσουμε στο πνεύμα αυτό της συνεργασίας και ελπίζω το τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι για το οποίο θα είμαστε υπερήφανοι γιατί πραγματικά είναι ένα σημαντικό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την κοινωνία. Σας ευχαριστώ κύριε Ματιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λούνατσεκ και χαιρόμαστε βεβαίως για την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι ήταν αξιόλογο το έργο των σκιωδών εισηγητών και όσον αφορά τη μα πολιτική ομάδα, όπω είπε και ο Μπέρτα Λίλη, το συζητήσαμε και τώρα θέλουμε να πούμε για το 2014 και για το 2016 ότι έχουμε κάποιε μικρέ επιφυλάξει ε, για το αν θα δώσουν το πράσινο φω. Ε, υπάρχουν πολλέ επιφυλάξει ε, στην ομάδα μα, τα συζητάμε τέλο πάντων, αλλά θα ήθελα να σα πω ε, και σε εσά και και στου άλλου συνεισηγητέ. Μπράβο για τι προσπάθειέ σα, τέλο πάντων, για αυτό το χάρτη πορεία που κατά την προσωπική μου άποψη είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό ε, και αυτό δεν είναι μόνο δική μου άποψη. Οπότε θα ήθελα να σα πω ότι εγώ πάντω θα ψηφίσω ε, όσο γίνεται πιο πολλέ από τι τροπολογίε που θα κρυφθούν στην Επιτροπή. Yes, thank you, Chair. I will join those who... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. λέει ε, κύριε κυρία Νιτφέλ και εγώ επομένω να πω μπράβο στους συζητητέ. Ε, βλέπουμε πόσο ευρεία είναι η συνένεση ε, στην Επιτροπή μας και εάν δεν διαφωνείτε έχουμε 14 κράτη-μέλη τα οποία έχουν τώρα προσυπογράψει την προσπάθεια αυτή για το χάρτη πορείας οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την αρνητική τη στάση και γι' αυτό και νομίζω ότι τη σήμερα μέρα θα πρέπει να δει η Επιτροπή ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο το μήνυμα από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε και τα μισά κρατημέλη επομένω και άρα θα πρέπει να κάνει το βήμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τελειώσει η θητεία τη. Αυτό ήθελα να πω. Πρόεδρος. To react right on the spot. Θέλετε τώρα ενθερμό να πείτε. Ναι, ναι, ναι, ήθελα να πω υπέρ τη Vivian ότι όταν τα 14 κράτη-μέλη προσυπέγραψαν ε, αυτή την, την, την, την, την έκκληση ε, ε, για να υπάρχει, ε, αυτός ο χάρτης πορείας, ε, τότε το κατέβασε αυτό σαν πρόταση στο Συμβούλιο η, η κυρία Ρέντινγκ, αλλά τα ίδια αυτά κράτη-μέλη ε, άλλα στο Συμβούλιο. Άρα θα πρέπει ε, να ξέρουν τη στάση τους. Και Κύριε Σιγιάνγκ, ευχαριστώ και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Λούνατσεκ για την έκθεσή τους και για τις ε, τροπολογίες, τις μόνες τροπολογίες που δεν συνυπέγραψα, αυτά αφορούν την ε, πολιτική εκπαίδευση και υγείας. Ε, και αυτό όχι επειδή διαφωνώ με την ουσία, αλλά για λόγους επικουρικότητας. Έτσι ώστε νομίζω το καλύτερο είναι η να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις εκθέσεις. Ε, επίσης, αν το θέλει ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν νομίζω πως μπορούμε πλέον να το αποφύγουμε και χαίρομαι για το ότι για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα θα ε, μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο. Σας ευχαριστώ, κύριος Μισελ. Όλα, όλα τα είπατε. Λοιπόν, θα πρέπει και εγώ απλώς να συγχαρώ την κυρία Λούνετσεκ για την εκθεσή της. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση. Όπως είπε και ο τελευταίος που έλεγε το λόγο, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα το οποίο στέλνουμε. Και άρα δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξει κάποιο είδους αντίδραση, κάποιο είδους απάντηση από πλευράς του Συμβουλίου και εγώ επίσης να σας πω ότι δεν μου αρέσει η τροπολογία 5. Τα είπε και ο Μάικλ Κάσμαν ότι τελικά πρόκειται για ε, κάτι το οποίο, πώς να το πούμε, ε, είναι, είναι, είναι μασκαρεμένο, δηλαδή δείχνει, δείχνει να είναι κάτι το θετικό, αλλά ουσιαστικά είναι το αντίθετο. Κατά διαβολικό τρόπο αποκρύπτει ε, ότι βάζει κάποιους φραγμούς εδώ και πέρα θρησκευτικής και λοιπά υφής και εγώ ως φιλελεύθερος Είμαι κατά, κατά τα άλλα δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσουμε όλα όσα ελέγχθησαν. Μπράβο στην κυρία Λούνιτσεκ για τα όσα έκανε. Ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ από ό,τι φαίνεται οι συνάδελφοι εκτιμούν ιδιαίτερα τη δουλειά σα, Έχετε το λόγο. Ναι, κάποια λόγια τελευταία. Ευχαριστώ όλους του συναδέλφους για τη στήριξή του και τον Λουί Μισελ για αυτά τα οποία είπε για την τροπολογία 5 αλλά όπως είπα και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Ματιέ που ξεκαθάρισαν πως ε, ελπίζω να έχουν περισσότερη στήριξη στην ομάδα τους με την τροπολογία αυτή. Δεν περίμενα τόσο υψηλό επίπεδο συνεργασίας και νομίζω πως κάτι κάνουμε όχι μόνο στο κοινοβούλιο αλλά όπως είπατε η Κομισιόν πλέον δεν μπορεί να αποφύγει το θέμα. Ελπίζουμε λοιπόν η επόμενη Κομισιόν να κάνει κάτι, άλλο για τα κράτη-μέλη. Τα 14 που συνυπέγραψαν φαντάζομαι στις χώρες όπου υπάρχουν συμμαχικές κυβερνήσεις όπως στη δική μου. Ξέρω έναν υπουργό που είναι υπέρ και υπέγραψε αλλά ο υπουργό Δικαιοσύνης δεν θα υπογράψει. Γι' αυτό μάλλον υπάρχει αυτό το θέμα στο Συμβούλιο κυρία ματιά φαντάζομαι γνωρίζετε ότι πάντοτε τελευταία λέξη τη λέει ο εισηγητής, αλλά αν θέλετε κάτι να προσθέσετε σε σχέση με αυτά που ακούσατε, στο λέει Μισελ θέλω να πω. Ότι για την τροπολογία 5 ξέχασα. Θα πρέπει να μιλήσω και να υπερισπιστώ τον συνάδελφο που συνέταξε την τροπολογία γιατί αυτό το οποίο θέλει να γίνει σεβαστή η ελευθερία της έκφρασης και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ακριβώς κάτι το υποκριτικό, κάτι που υποκρύπτει κάτι άλλο. Δεν συμφωνώ. Αυτό ήθελα να πω. Μισελ. Ναι, ναι. Βεβαίω και καταλαβαίνω τι θέλει να πει η κυρία Ματιού. Καταλαβαίνω ότι θέλει να επιδείξει αλληλεγγύη προς κάποιον πολιτική της ομάδα. Και καταλαβαίνω ότι σας φέρνει αμηχανία αυτή η τροπολογία. Αλλά δεν, δεν, δεν αλλάζω ούτε μια κεραία, ούτε ένα ιότα από όσα είπα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι υποκρύπτεται κάποια άλλη πρόθεση πίσω από αυτή την τροπολογία και τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκει σύμφωνο σε σχέση με όσα πρεσβεύω για τη δημοκρατία και για τον σεβασμό των ε, ανθρωπίνων επιλογών. Ωραία, θα περάσει από ψηφορία και γιατί είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο γιατί έτσι ανοίγεται μια κερκόπορτα ή μια ερμηνεία η οποία θα είναι πάρα πολύ ευρία ευρετάτη, για ό,τι να είναι. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι δόκιμη. Τέλο ο καθένα έχει την άποψή του. Oh, voilà. Ε, Madame Lunacek, would you like to add anything? Nothing else. θέλετε Όχι, ευχαριστώ. Ε, εντάξει, έκλεισε επομένω το θέμα και προχωρούμε. Πάμε ή στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι το 7. Πολύ σημαντικό. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για αυτό το σημείο αφορά τον συνάδελφο κύριο Γιακολίνο που είναι ο εισηγητή, αλλά δεν είναι εδώ. Πώς, πού είναι, έρχεται. Α, ναι, είμαι σίγουρο είμαι σίγουρος ότι έρχεται. Έρχεται, έρχεται. Επομένως, αν την καλοσύνη, ας δείξουμε υπομονή για λίγα λεπτά να περιμένουμε να έρθει ο κ. Γιάκουλον και να κάνει την εισήγησή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. So thank you. Thank you Ευχαριστώ για την υπομονή που επιδείξατε, λέει ο Πρόεδρος. Και για τη συνεργασία επίσης. Οπότε ήρθε ο συνάδελφος κύριος Γιακολίνο που βρίσκεται εδώ ή στο Προεδρείο για να εισηγηθεί το θέμα του που αφορά την ε, διάμεση έκθεση για την Ευρωπαϊκή Σαγγελία. Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Στις 17 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της, το σχέδιο κανονισμού όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επιτέλους, γιατί πρόκειται για την ίδια τη συνθήκη της Λισαβόνας συγκεκριμένα, η νομική βάση είναι το άρθρο 86 της Συνήθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το θέμα αυτό πρόκειται για μια νομική επανάσταση. Πρόκειται για μια σειρά ζητημάτων τα οποία ήταν στην σφαίρα της ε, κυβερνητικής να μεταξύ κρατών μελών και όλα αυτά Ε, έπρεπε να αναχθούν στο του ευρωπαϊκού δικαίου και πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης η συνήθις νομοπαρασκευαστική διαδικασία Ε, Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και μία από τις εξαιρέσεις είναι το συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 86. Δεν υπάρχει επομένω στη συνήθεια νομοθετική διαδικασία την συναπόφαση. Όμω, όμως, σύμφωνα με την ε, διατύπωση του 86, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί, να ληφθεί υπόψη η άποψή του και θα πρέπει να δώσει το πράσινο φω, τη συνένεση, την έγκριση για το τελικό κείμενο όσον αφορά αυτόν τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θεσμικό βήμα προς τα Γι' αυτό αφορά έρευνες, ανακρίσεις, άσκηση ποινική δίωξης προς και κατά εκείνων οι οποίοι ενεργούν κατά των συμφερόντων της ε, ενόμου τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συμφερόντων της και τελικά πρόκειται για μια διεύρυνση των ε, κοινωτικών αρμοδιοτήτων σε σχέση με την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος συγκεκριμένα για τα εγκλήματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 83 της ε, Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι συντονιστές μας αποφάσισαν να γνωμοδοτήσουν. Οπότε και αποφασίστηκε να ανατεθεί στο Κυριακό αυτή η διαμεσή έκθεση, ο οποίο βρίσκεται εδώ για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Το κείμενο, από ό,τι γνωρίζω, διατίθεται ή στα Ιταλικά πώ το παρόν. Αλλά υπάρχει μετάφραση στα Αγγλικά. Οπότε ακούσουμε με είχε να μας πει ο Γιακολίνο για το σχέδιο έκθεσης και στη συνέχεια να συζητήσουμε το κείμενο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπατε σαφέστατα στη σύντομη αλλά πολύ ακριβή ανακεφαλαίωση τι θέση θα έχει αυτό το νομοθέτημα στην οικοδόμηση του αρχιτεκτονήματος της Ευρωπαϊκής Θεσμικής Διοργάνωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον προπολογισμό που αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες, σημαντικοί πόροι, οι οποίοι πρέπει να προστατεύονται καλύτερα. Μιλάμε για, τις, για τα μεγάλα έργα για τον πολιτισμό που σαφώς χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό το νομοθετικό ζήτημα ε, καλύφθηκε μαζί με τη Eurojust. Και ένα άλλο θέμα που αφορά τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα ντοσχέ το οποίο βάσει του άρθρου 86 της συνθήκης θα οδηγούσε στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιας ε, ελαφριάς ε, και ευέλικτης και αποτελεσματικής εισαγγελία που θα βρισκόταν υπό την επίβλεψη των εθνικών κοινοβουλίων. Όπως τα ξέρετε, 14 εθνικά κοινοβούλια τοποθετήθηκαν αρνητικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτός είναι ένας από τους λόγους που στις 16 Δεκεμβρίου θα μιλήσουμε με την κυρία Ρέντινγκ για το θέμα αυτό και συνολικά για το πακέτο δικαιοσύνη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των προτάσεων εδώ με τους συντονιστές. Είχαμε μια συζήτηση κάποιες φορές εντατική αλλά συνήθως επικοδομητική. Τους ευχαριστώ λοιπόν αυτής εξ αρχής διότι και βάσει γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας για συγκεκριμένα στοιχεία, για τη νομική βάση, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ξεκαθαρίσαμε κάποια θέματα. Θεωρήσαμε πάντως εύστοχο για το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτό το τελευταίο τμήμα θητείας που του μένει να αποφανθεί το Κοινοβούλιο για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που θα μπορούσε να τα αξιολογήσει το Κοινοβούλιο θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται με το φυσικό δικαστήματο, με τα συμπληρωματικά αδικήματα. Εδώ ζητούμε συγκεκριμένη αναθεώρηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε ότι παρόλο που είναι βοηθητικός ο ρόλος μας στην εξέταση του θέματος αυτού, πρέπει να παρακολουθήσουμε το θέμα και να υπάρξει συμφωνία επί της ουσίας στα πιο σημαντικά περιεχόμενα. Για τα άρθρα 27, 28 και 29 τοποθετηθήκαμε, ζητούμε την προστασία των δικαιωμάτων κατηγορουμένου, διαδικαστικές δικονομικές διασφαλίσεις, επίσης η εισαγγελία να αποτελείται από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών, δηλαδή να υπάρχει κύρος και συγκεκριμένες βάσεις. Και βεβαίως θα πρέπει να καθοριστεί και η σχέση με την Όλαφ, της εισαγγελία δηλαδή και της Όλαφ. Αυτά είναι στοιχεία που θα τα αναπτύξουμε και σε άλλες εκθέσεις, αλλά εν μέρη και σε αυτήν. Επίσης, εντοπίσαμε τον προσωρινό χαρακτήρα της έκθεση αυτή. θα μπορούσαν να ακολουθήσουν κι άλλες, προκειμένου να ζητήσουμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τη σκοπιά του Ευρωκοινοβουλίου. Περνάω στα συμπεράσματα. Ζητούμε από το Συμβούλιο να υλοποιήσει τον πίνακα, τον χάρτη πορείας για τις ε, διαδικασίες της ποινική ολοκλήρωσης, ε, και με μέτρα για την έρευνα που θα πρέπει να διέπονται από τις σχετικές αρχές για τη λειτουργία της εισαγγελίας. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ε, ευρωπαϊκό ποινικό χώρο, διαφυλάσσοντας βεβαίως τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, πρέπει να προχωρήσουμε. Είμαι πεπισμένος και ολοκληρώνω ότι οι ενέργειες αυτές μπορούν να προχωρήσουν βάσει ενός χρονοδιαγράμματος που έχουμε καταστρώσει την, ε, από κοινού με τη γραμματεία αλλά και με την ευκαιρία των συναντήσεων των σκιωδών αφού εξέφρασαν τις εκτιμήσεις τους οι συνάδελφοι βάσει των ε, όσων επιθυμούν οι πολιτικές ομάδες. Ελπίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα μέσα στη χρονιά να έχουμε και την ομάδα της Ιδης Υπηρεσίας η οποία εργάζεται δυτικά προς αυτό το σκοπό. Η ημερομηνία της 17ης Ιανουαρίου έχει προβλεφθεί για τις τροπολογίες, 30 Ιανουαρίου για την εξέταση των τροπολογιών, 12 Φεβρουαρίου θα μπορούσε να προβλεφθεί η ψηφοφορία στην ΛΥΜΠΕ για να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Τον Απρίλιο, όπως ξέρετε, τα μόνα θέματα που μπορούν να συζητηθούν και να ψηφιστούν στην Ολομέλεια είναι τα νομοθετικά. Είναι λοιπόν μια υπόθεση εργασίας αυτή. Θα χρειαστεί στήριξη των σχεδόν εισηγητών, αλλά πιστεύω ότι δεν θα παραλείψουν να βοηθήσουν, όπως εξυπηρέτησαν ως τώρα όλοι οι συνεργάτες, για να πετύχουμε ένα σκοπό που είχαμε προκαθορίσει. Θα σταματήσω εδώ πρόεδρε θυμίζοντας ότι είμαστε στη διάθεσή σας, όπως και η Γραμματεία της Επιτροπής που εργάζεται πολύ συγκεκριμένα για το θέμα αυτό. E Ας ακούσουμε λοιπόν διαφορετικές απόψεις για να δούμε πώς μπορούμε να τις συνθέσουμε και το Ευρωκοινοβούλιο να προσφέρει τη δική του οπτική γωνία σε αυτή τη ε, δράση του Συμβουλίου μεγάλη στρατηγική αξία το θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που δεν είναι καθόλου απλό. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε του σκιαδεσίτε. Θα ακούσουμε την κυρία Τσίπερ πρώτα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνο για τη δουλειά που έχει κάνει, γιατί νομίζω πως όλες οι ομάδες υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά που πρέπει να ξεκαθαρίσουν και επειδή αναφέρθηκαν κάποια πράγματα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο-τρία βασικά ζητήματα. Ήδη αναφέρθηκε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να πάει σε μια διαδικασία σύμφωνης γνώμης, κάτι το οποίο βεβαίως δεν αμφισβητείται. Επίσης, ε, πολλοί σκιώδης αγγελής είχαν ενοχληθεί γιατί η πρόταση της Κομισιόν είναι πάρα πολύ λεπτομερής και υπήρχαν δύο σημεία κριτική. Το ένα είναι πως βεβαίως ο Ευρωπαίος εισαγγελέας ε, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά του αποτελεσματικά. Οπότε χρειάζεται αρμοδιότητες και να μπορεί να ξεκινήσει έρευνες, αλλά βεβαίως πάντα παραπέμπουμε στις εθνικές διαδικασίες οι οποίες ε, και βεβαίως σε διαδικασία προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των δικονομικών δικαιωμάτων ε, ευρωπαϊκών, αλλά στην πρόταση γίνεται λόγος και για δικονομικά δικαιώματα που θα προκύψουν, όπου ελπίζω πράγματι να πάμε πέρα από αυτά τα οποία αναφέρονται στο κείμενο. Και έτσι υπήρχε και θα υπάρξει μια συζήτηση για αυτό το θέμα γιατί η ποινική δίωξη βεβαίω ε, προχωράει αφενός αλλά πρέπει και να προστατεύονται και τα δικαιώματα των κατηγορουμένων στο ίδιο επίπεδο. Γι' αυτό είμαστε υπέρ την πρόταση, της πρότασης ε, για έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα, αλλά βεβαίως είπαμε πως ε, η εισαγγελία αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί κατά έναν τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματική ε, και να λειτουργεί χωρίς σοβαρά προβλήματα. Να σας υπενθυμίσω πως μιλάμε ήδη για αλλαγές σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο έχει οδηγήσει σε προβλήματα τα τελευταία χρόνια και βεβαίως δεν θέλουμε κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτό. Γι' αυτό έχουμε κάποιες ερωτήσεις ακόμα που υποβάλαμε στην νομική υπηρεσία και ελπίζουμε να λάβουμε απάντηση φέτος. Σημαντικό είναι λοιπόν να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση της Κομισιόν για τη διαδικασία της πράσινης κάρτας είναι ένα σημαντικό ζήτημα και βέβαια έχουμε και το θέμα των συγκεκριμένων ορισμών. Τι είναι και βεβαίως τι γίνεται με την απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ειδικά για αυτό το τελευταίο Πρόκειται για απάτη εις βάρος των συμφερόντων όλων των ε, φορολογούμενων, των πολιτών μας. Οπότε θα πρέπει να επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς το συμφέρον των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω πως έχουμε ψηφοφορία στις 10.30 και μετά βεβαίως ε, θα έχουμε και τη συζήτηση. Οπότε παρακαλώ να μείνετε στην ουσία για να προλάβουμε την ψηφοφορία στις 10.30. Κυρία Βίλεμ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τη γραμματεία. Δεν έχω πολλά σχόλια επί της ουσίας του σχεδίου έκθεσης. τη στηρίζουμε. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να ε, συζητήσουμε κάποιες άλλες πτυχές που έχουν μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δυστυχώς έχω την αίσθηση πως μέχρι στιγμής έχουμε στείλει λάθος μήνυμα. Δηλαδή, ε, αν έχει αντίρρηση ένα εθνικό κοινοβούλιο, δεν σημαίνει πως συμφωνεί με την απάτη βάρους των οικονομικών σφαίρων της Ένωσης, έτσι. Απλά... Ε, δεν συμφωνεί με όλες τις πτυχές. Επίσης, εδώ πέρα νομίζω συμφωνούμε με όλες τις πτυχές και τον εισηγητή πως ναι, θέλουμε αυτό το οποίο προβλέπει το άρθρο 86 της συνθήκης, όμως υπάρχουν και άλλες πτυχές. Ε, γιατί το κοινοβούλιο εδώ πέρα βρίσκεται απλά σε μια, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας σύμφωνης γνώμης. Αυτό ορίζει το άρθρο 86. Όμως τι έκανε η Κομισιόν. Πήγε πέρα από τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 86 και ανέφερε επίσης ε, ζητήματα που αφορούν τα διαδικαστικά δικαιώματα των κατηγορουμένων, ε, τεκμήριο αθωότητας, ε, νέμπις in idem και τα λοιπά. Και σε όλες αυτές τις πτυχές κατά κανόνα έτσι κάνει το κοινοβούλιο. Κατά κανόνα είναι στην διαδικασία της συναπόφασης. Εμείς θεωρούμε λοιπόν πως η Κομισιόν δεν σεβάστηκε το άρθρο 86. Γι' αυτό ζητήσαμε τη γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας, αλλά και της υπηρεσίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά δεν είναι παράπλευρα, έτσι. Είναι πολύ σημαντικά, γιατί το να στερηθεί το κοινοβούλιο το συνταγματικό του δικαίωμα να συναποφασίζει και να συνομοθετεί είναι κάτι το πολύ σοβαρό κατά κανένα τρόπο, επειδή αναφέρατε το άρθρο 83, 83 ε, ε, και την δυνατότητα που έχει το ε, όργανο αυτό να μεταβληθεί σε εισαγγελέα που θα ασχολείται και με άλλα εγκλήματα. Όχι. Είναι de Generalis το άρθρο 82 και de Specialis το άρθρο 83, 86. Οπότε να δούμε το άρθρο 86 πρέπει να δεχτούμε πως το Κοινοβούλιο είναι αυτή τη στιγμή σε διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Το 83 είναι συναπόφαση. Αν λοιπόν θέλουμε μια γενική ευρωπαϊκή εισαγγελία κάποια στιγμή πρέπει να ε, εφεύρουμε κάτι νέο και όχι να μετασχηματιστεί αυτό το θεσμικό όργανο. Δεν ξέρω, μπορεί να σας φαίνονται πολύ νομικίστικα αυτά, αλλά όχι. Ε, σχετίζονται με τα δικαιώματα των εκπροσώπων των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία υπόθηκαν και άρα θα μείνω σε κάποια θέματα Όσον αφορά την ουσία του σχεδίου έκθεση, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι όλες οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει ε, για όλες τις αποφάσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί ε, έφεση, ειδικά στο άρθρο 13 όπου υπάρχει εξαίρεση από την ε, δυνατότητα επανεξέτασης ε, της υπόθεσης. Δεν νομίζω πως είναι σωστό αυτό. Επίσης και το θέμα της δικαιοδοσίας και το ποιο δικαστήριο επιλέγεται. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, προσφυγής ε, και έφεσης. Το άλλο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι πως πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως δεν πρέπει να επιλέγει σε ποια δικαιοδοσία θα πάει κάποιος για να μην παρακάμπτει δηλαδή τις διαδικασίες κρατών μελών οπότε πρέπει να ενισχυθεί αυτό το κομμάτι. Νομίζω πως όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα και τις αρχές ε, όσον αφορά τη συλλογή αποδεκτικών στοιχείων τα δικαιώματα της υπεράσπισης. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα και είναι και αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πως τα δικονομικά δικαιώματα δεν επιτρέπεται να υπονομεύονται όσον αφορά το επίπεδο προστασίας ε, θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Ε, δεν πρέπει λοιπόν όπως είπα να υπάρχει κάποια μείωση ε, της ε, προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη και θα έλεγα μάλιστα ε, επειδή σε 20 λεπτά ψηφίζουμε για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας για μια πάρα πολύ ευαίσθητη ευαίσθητο συμβιβασμό και λεπτό, νομίζω πως αυτό πρέπει να φαίνεται και στο πώς αντιμετωπίζουμε τις ε, διάφορες ρήτρες ε, προστασίας, τις δικλείδες ασφαλείας και πρέπει νομίζω να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τέλος. Όσον αφορά την συζήτησή μας και τα προβλήματα με τον Όλαφ. Πλήρης ανεξαρτησία δεν σημαίνει πως στο τέλος η πολιτική ευθύνη για παραβιάσεις θεμελιώδης ε, από τα θεσμικά όργανα να είναι στα ίδια τα θεσμικά όργανα. Όχι. Η ευθύνη ανήκει στην Κομισιόν που έχει μια πολιτική ευθύνη για τα λάθη που μπορεί να γίνουν από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει την ευκαιρία να δείτε το τι γίνεται με τον πολιτικά υπεύθυνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φως. Ε, γρήγορα παρακαλώ γιατί έχουμε και ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ήθελα να υπενθυμίσω το γιατί είναι σημαντικό το να σκεφτούμε αυτή τη μελλοντική δομή και αυτό το συζητήσαμε και χτες στο πλαίσιο της συνάντησης των σκιωδών για την Eurojust και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Eurojust σχετίζονται και επιπλέον βεβαίως υπάρχουν και άλλα θεσμικά όργανα όπως ο Όλαφ, η Europol οπότε πρέπει να σκεφτούμε το πώς γενικά θα κάνουμε κάτι σε αυτόν τον τομέα και όσον αφορά τις διπλές αρμοδιότητες αυτές πρέπει να αποφευχθούν αλλά πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με την συνεργασία με την εισαγγελία, με την αστυνομία, ποιες είναι οι αρμοδιότητες των δικαστηρίων, τι γίνεται με την ποινική δικονομία Μετά αυτό το οποίο αναφέρθηκε για κάποιες αρχές ευρωπαϊκές όπως το in Idem ε, και διάφορα άλλα θέματα και επίσης η ιδέα της ε, νομικής ε, αρρωγής πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πως όλο αυτό το θέμα Πώ ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το θέμα των δικονομικών δικαιωμάτων και άρα χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο. Κύριε Ντεγιόγκ, σύντομα παρακαλώ, γιατί έχουμε να ακούσουμε και την Κομισιόν και τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα δεν συμφωνώ με αυτούς που είπαν πως υπάρχει συνένεση για την ανάγκη ε, Ευρωπαίου εισαγγελέα Νομίζω πως έχει ξεκαθαρίσει πως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες τις οποίες δεν ερεύνησε η, δυνατό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως να υπάρχει ένας Ευρωπαίος, ε, ένας με συγχωρείτε εθνικός συνομιλητής ε, σε κάθε χώρα αναμένω και εγώ αυτό το οποίο είπε η κυρία Βέμπερ, την ε, νομική γνωμοδότηση για τις αρμοδιότητες, αλλά ακούω πως το Συμβούλιο τον Μάρτι που έρχεται θα αποφασίσει για μια διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας, εάν περάσει κάτι τέτοια και κάποια κράτη-μέλη ε, περάσουν σε, ένα, Ευρωπαίο εισαγγελέα, και κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν περάσουν σε αυτό το καθεστώς. Τι σημαίνει αυτό για τη Eurojust, τι σημαίνει για τον Όλαφ. Ε, πρέπει να τα δούμε αυτά. Είναι πολύ ουσιαστικά ερωτήματα. Είναι για την άποψη, κατά την άποψη της ομάδας μας εξαιρετική σημασία. Μάλιστα. Ας ακούσουμε τώρα την Κομισιόν. Ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελε να παρέμβει. Θέλετε το λόγο, υπάρχει πρόσωπος της Επιτροπής. I was looking for you. Mr. Chairman, thank... Ναι, ναι, εσάς. Εσάς Ευχαριστούμε Πρόεδρε και χαιρετίζουμε αυτήν την ε, τόσο μεστή έκθεση του κυρίου Γιακολίνα. Συμπαθάτε με μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Έτσι γίνεται συνήθω πριν την ψηφοφορία. Οπότε παρακαλώ εσεί που έρχεστε στην αίθουσα κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να ακούσουμε την Επιτροπή αλλά και το, τον εισηγητή που θα πει τελευταία λέξη. Ε, ευχαριστούμε για αυτή την ολοκληρωμένη έκθεση του Ιακολίνα, κύριε Πρόεδρε, και θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα θετικό βήμα πρόοδο και όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα έχει προβεί στην έκδοση ανακοινώσεως όσον αφορά ε, τις ε, αιτιολογημένες ε, γνωμοδοτήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στη συζήτηση έχουν θυγεί αυτές τις γνωμοδοτήσεις, έχουμε και τις ε, διοργανωτές που θα ακολουθήσουν και εμείς έχουμε δεσμευτεί να λάβουμε υπόψη όσο έχουν πει τα Εθνικά Κοινοβούλια κατά εκείνες τι ε, διαπραγματεύσει, οι οποίε είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν κάποια συνέχεια. Τώρα θα ήθελα κάτι απλώ να σα αναφέρω όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα στην πρότασή μα. Νομίζουμε ότι θα πρέπει το κείμενο να είναι ε, να έχει κάποια ιστορική συνοχή. Άρα θα πρέπει να καλύψουμε τα δικονομικά δικαιώματα, ε, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί σε άλλο κείμενο. Θα πρέπει σε αυτό το κείμενο να ρυθμιστεί η ισότιμη μεταχείριση δικονομικών δικαιωμάτων, αλλά και των λεπτομεριών ε, των εισαγγελικών ενεργειών, έρευνών κλπ και έτσι να υπάρχει ε, μια εισαγγελική υπηρεσία η οποία να είναι ανεξάρτητη, αμερόληπτη και αποτελεσματική. Θα σε ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Γιακολίνο για να κλείσει το θέμα ως εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χρήσιμες όλες οι συνεισφορές των ε, σκιωδών κατά την εκπόνηση της έκθεσης και ήταν χρήσιμες και οι σημερινές σας ενδείξεις. Βεβαίω θα επιδιώξουμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει παρουσία σε όλα τα κρατημέλη, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό σκέλος της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Το ευρώ αφορά 18 ε, χώρες πλέον και μια είναι αγορά που απλώνεται σε 30 κράτη. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα να διορθωθεί βάσει των συνεισφορών των σκιωδών και άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μα μάλλον, που θα τοποθετηθούν για τα θέματα αυτά. Ε, δεν θέλουμε η έκθεση να είναι άκρο λεπτομεριακή. απλώ η δική μα οπτική γωνία που ελπίζουμε ότι θα απασχολήσει μέχρι, θα φτάσει στα χέρια των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων στο Μάρτιο του 2013 14 μάλλον, θα ληφθεί επαρκώς υπόψη ώστε να βελτιωθεί ένα κείμενο το οποίο καλό θα ήταν να συνδυαστεί και με άλλα νομοθετικά κείμενα του ευρύτερου πακέτου δικαιοσύνης. Θα ήθελα λοιπόν οι υπόλοιποι εισηγητέ που είναι υπεύθυνοι για τα υπόλοιπα ντοσιά, τα υπόλοιπα θέματα, να τα προωθήσουν με την ίδια σύνεση, την ίδια επιμέλεια και την ίδια σχολαστικότητα όπως έχουν κάνει ως τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμεί, κύριε Γιακολίνο. Ε, έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση, οπότε απλώ να σα υπενθυμίσω ότι η υποβολή των τροπολογιών έχει όριο προθεσμία και τελική τέλο πάντων την 17η πρώτου την μεσημβρία του, του χρόνου. Οπότε, εδώ προχωρούμε στι ε, ψηφοφορίε Είστε έτοιμοι. Βεβαίω και θα πρέπει να έχετε έτοιμη την ε, κάρτα τη ηλεκτρικής ε, ψηφοφορία. Όποιο δεν την έχει, α στείλει να του τη φέρουν. Και προχωρημένο με το σημείο παριθμών 8 που αφορά την εφαρμογή των στρατηγικών για του Ρωμά. Πρόκειται να υποβληθεί αυτό το κείμενο στην Ολομέλεια από πλευρά τη Επιτροπή μα κατόπιν των αντιστοίχων προφορικών ερωτήσεων προ Συμβούλιο και Κομισιόν για το ίδιο θέμα. Οπότε τώρα θα αρχίσουμε. Αρχίζουμε. Those in favor. Όλες οι τροπολογίε από α μέχρι χ. όλε μαζί υπέρ, κατά, αποχές ψηφίζουμε. W, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, ωραία. Ε, τώρα εδώ καλύπτονται πάρα πολλά θέματα και φτάνουμε μέχρι το 153 και είναι υπέρ είναι κατά αποχές Και μετά είμαστε στο 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν σε το αποτέλεσμα έλεγχος. 156 έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Για να δούμε τι αποτέλεσμα έχουμε. Αγωγιακή η ψηφοφορία. Χαιρετούμε και εσείς ψηφίσατε. So it's 20 plus, 19 against. It's been adopted. Now, 155. 155. Όχι, όχι. Αυτή καταπίπτει. Πάμε τότε στο 158. Τι είναι υπέρ. Κατά. Απογείες. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Καλά, τότε να θεωρήσουμε ότι απορρίπτεται. Ψηφίζουμε. Εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται. Τέλος να ξαναψηφίζουμε. Σηκώστε καλά τα χέρια. Πέρας.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 18 καλύπτεται από την ε, συμβαστική α, άρα πάμε στο 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 20, όχι θα κάνουμε έλεγχο για την ψηφορία επί της 19. Ψηφίζουμε. Πέρας. Οριακό το αποτέλεσμα πάντως απορρίπτεται. Πάμε στο 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχο για το 26 κάνω. Πέρας. 21-22 και πάλι. Α, αυτή τη φορά εσείς νικάτε. ωριακά, αλλά Νικήσατε. 35. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 38. Κατά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 Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πέρας. 22-21 και πάλι. Άρα περίφθη. Κάνουμε τώρα την τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Σαράντα. Ένα. Δύο εποχές. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Γιάννη. Και τώρα θα ψηφίσουμε την εκθέση Νούνου Μέλου. Σχέδιο εκθέσεω για, την, για το ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνα σε ποινικές υποθέσει. Voting Melos Report, European Investigation Order. Are you ready? Είστε έτοιμοι? Τροπολογία 200, υπέρ. Ναι. Ναι, ναι, συμβιβαστικό κείμενο. Τροπολογία 200. Ναι. Υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε στα άρθρα. Όλα αυτά τα γλιτώνουμε. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Σαράντα δύο υπέρ. Μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια κύριε Μέλου. Α, αυτός ήταν συμβιβασμός με το Ευρωπαϊκό Έντελμα Έρευνα. Έχετε το λόγο. Σύντομα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεισέφεραν τους οι εισηγητές για τη βοήθειά τους τον Γιώζεφ Βάιντα Χόλτσερ, τον κύριο Βανσέτα, την Βαρόνι Λάτφορντ, την κύριο Άλμπρεχτ, Τίμωθη και τον κύριο Κορνέλης, γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρναμε και έτσι καταφέραμε να βελτιώσουμε το έργο αυτό. Άσχημα νέα λοιπόν για τους εγκληματίες και θα τους διώκουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Μελού για την έκθεσή σας, για την παρουσίαση και για τη συμβαστική σας πρόταση, γιατί οπωσδήποτε μας βοηθάνε αυτά με τη ρησφοφορία. Περνάμε σημείο 4. η κατάσταση των διοργανικών διαπραγματεύσεων σε νομοθετικές διαδικασίες που έχουν το αποτέλεσμα ε, που το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Colleagues, little silence in the room. Ησυχία παρακαλώ συνάδελφοι. ησυχία. Είστε έτοιμοι. Όπως έλεγα. Έχουμε να ακούσουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της οδηγίας των ε, κατασχέσεων. Κυρία Μακοβέη, συγγήτρια, θα μας ενημερώσει τώρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, πραγματί τελειώσαμε. Είχαμε την τελευταία φάση την προηγούμενη εβδομάδα και η Κορεπέρ ψήφισε το κείμενο πριν από δύο ημέρες. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των σκιωδών από τους σοσιαλδημοκράτες, ε, την Άλντε και την Γκούε, οι παρόντες έλαβαν μέρος στις διαπραγματεύσεις και σύντομα να σας πω για τις εκτεταμένες ε, κατασχέσεις είχαμε αρκετά πράγματα Δηλαδή οι περιπτώσεις που καλύπτονται είναι δωροδοκία και δωροληψία και στο δημόσιο τομέα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους υπαλλήλους της Ένωσης, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με οικονομικό όφελος. Προσθέσαμε και το έγκλημα και την παιδική πορνογραφία. Επίσης υπάρχει μια ρήτρα για αναθεώρηση από την Κομισιόν για να επεκτείνει τον κατάλογο αυτών των ε, αδικημάτων για να προσαρμόζεται στις τάσεις του οργανωμένου εγκλήματος για κατασχέσεις από τρίτους ε, ισχυρές τρίτων ε, όταν θα έπρεπε όφυλα να γνωρίζουν πως ήρθε προϊόντα εγκλήματος, ε, όταν κάτι δηλαδή πωλείται και αγοράζεται κάτω από την εμπορική τιμή θα πρέπει να είναι δυνατή η κατάσχεση ισχυρά τρίτη. Και όταν μιλάμε η δυνατότητα να γίνεται αυτό και εμέσως. Όσον αφορά τις ρήτρες ασφαλείας, ε, ενισχύσαμε το άρθρο αυτό, μιλάμε για δίκη, δίκη, ενημέρωση βεβαίως για τους λόγους για τους οποίους γίνεται κατάσχεση ή ε, ε, δέσμευση. Μετά έχουμε το δικαίωμα της πρόσβασης βεβαίω δικηγόρο και τα δικαιώματα των θυμάτων. Επίσης η χρήση ε, των ε, κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων και επιτρέπεται, ενθαρρύνονται μάλιστα να τα χρησιμοποιήσουν ε, προς το κοινό συμφέρον. Θα ήθελα επίσης να αφαιρθώ στα της κατάσχεσης το οποίο μιλάμε για κατάσχεση ε, χωρίς ε, καταδίκη δεν υπάρχει στο κείμενο καθεαυτό. Τα κράτη-μέλη ε, πλην ενός δεν ήθελαν να δεχτούν την περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή της δίκης ε, να αιτιολογεί την κατάσχεση αλλά συμφώνησαν ε, στην περίπτωση ασθένειας και φυγής από τη χώρα. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν. Δηλαδή σε περίπτωση στην οποία κάποιος ε, είναι ασθενής και δεν μπορεί να δικαστεί ή έφυγε από τη χώρα, εάν θεωρηθεί πως τα στοιχεία θα οδηγούσαν σε καταδίκη. Ένα προσωπικό σχόλιο αλλά εδώ πέρα συμφωνούν και οι σκιοδεσηγητές από την άλλη και τους σοσιαλδημοκράτες. Είναι πολύ εύκολο για τα δίκτυα αυτά να βάλουν όλα αυτά τα αγαθά στο όνομα κάποιου άλλου και μετά αυτός να βρεθεί δολοφονημένος. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ε, δεν το δέχονταν αυτό τα κρατη και μετά περνάμε Βεβαίω και στην κατάσχεση μετά από δικαστική απόφαση, μετά από καταδίκη. Επίσης τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να δώσουν περαιτέρω και συγκομισιών όσον αφορά το τις ε, κατασχέσεις και δεσμεύσεις ε, και βεβαίως έχουμε μια κοινή δήλωση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και ζητάμε από την Κομισιό να αναλύσει το στομότερο δυνατόν την κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών, τα πιθανά ωφέλη περαιτέρω κοινών κανόνων για κατάσχεση ε, περιουσίας που είναι προϊόν εγκλήματος. και σε σχέση με την καταδίκη ατόμων για τι δραστηριότητε αυτέ. Όπω ακούσαμε, τη Ιρλανδική Προεδρία, η Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού είναι συνήθι πρακτική αυτά. Με αποτελέσματα Ναι, κάποιοι, κάποιοι, κάποιοι από εσά. Απαντάει η εισηγήτρια σε κάποια σχόλια εκτό μικροφώνου. Ε, κοιτάξτε, ε, εκεί στα ορεινά της αιθούς λίγο σεβασμό παρακαλώ στη, στη βουλευτή που έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα έχουμε αυτή την κοινή δήλωση Κομισιόν και Κοινοβουλίου για να ε, εξεταστεί η δυνατότητα κατάσχεσης ε, προϊόντων εγκλήματος ακόμα και χωρίς καταδίκη. Αυτό συμβαίνει στην Ιταλία, ε, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και είναι, ε, χρησιμοποιείται επιτυχώς. Αυτά λοιπόν και αναμένουμε και τις μελλοντικές εξελίξεις. Βεβαίως πρέπει να πω πως ευχαριστώ τον, την κυρία Μπορσελίνο και τη Σόνια Αλφανό δεν εδώ και τους υπόλοιπους κοιοδεσίγητες για την ε, συνεισφορά τους ε, και θέλω να τονίσω πως η Λιθουανική Προεδρία πραγματικά το προωθούσε αυτό το ζήτημα ευχαριστώ σας ευχαριστούμε κυρία Μακοβεή έχει σημασία αυτό πράγματι πλησιάζουμε στο τέλος της μας Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διεκπαιρεώσουμε αυτά τα οποία ακόμα εγκρεμούν και αυτό αφορά και τα ζητήματα ε, ποινικού δικαίου, δηλαδή για αυτές τις ε, κατασχέσεις ε, δημεύσεις, για την ποινική δικονομία κλπ. κλπ. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπήρχε αυτή η συμφωνία για τα ζήτημα μας είπε η κυρία Μακοβέ, την οποία και την ευχαριστούμε μας ενημέρωσε και τώρα αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι το πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη. Ε, αν δεν έχετε άλλε παρατηρήσει, κανεί δεν έχει ζητήσει το λόγο. Αν κάποιο άλλο δεν θέλει το λόγο. Α, κύριε Μπορσελίνο, εσεί θέλετε το λόγο. Ήμουν ό,τι εισηγήτρια και πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Μακοβαέ για τη δυσχερέστατη και περιπλοκότατη εργασία που πραγματοποίησε του τελευταίους μήνες. Υπάρχει μια σχετική απογοήτευση γιατί τα σημεία που τόνισε και η κυρία Μακοβέη δεν καταφέραμε να τα φέρουμε εις πέρας. Είμαι βέβαιη ότι η δίμευση σε περίπτωση θανάτου θα ήταν μια, ε, ένα μεγάλο βήμα πρόοδου γιατί η κληρονομιά θα ήταν παράνομη σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι μόνο αυτός που συσσόρευσε μια περιουσία αλλά η κληρονομιά γίνεται παράνομη εφόσον ο ιδιοκτήτης έχει πεθάνει. Μου φαίνεται ότι είναι κάτι που πραγματικά είναι μια δυναμία. Αλλά καταφέραμε άλλα σημαντικά και κάτι είναι και αυτό. Αποδεχτήκαμε τουλάχιστον αυτή τη συμβαστική πρόταση. Τα θέλαμε σίγουρα περισσότερα, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα. Ένα σημαντικό βήμα, μικρό ή μεγάλο, αλλά είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ορσελίνο, για όσα είπατε. Ως σκιώδης εισηγήτρια. Κάποιο άλλο βουλευτή θέλει να πει κάτι άλλο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Α, ο κύριο Ντεγιόνγκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύσκολες ήταν αυτέ οι διαπραγματεύσεις και ευχαριστούμε την κυρία Μακοβέ για όσα έκανε. Κάπω ε, διαφορετικά τα βλέπουμε εμεί από ό,τι άλλε πολιτικέ ομάδε γιατί νομίζουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα ε, αντικατοπτρίζει περισσότερο την αρχική μα ε, τοποθέτηση ω ομάδα. Τώρα συζητήσαμε την έκθεση, οπότε ε, εμεί χαιρόμαστε και για το ένα αποτέλεσμα, αλλά και για το τι είδου αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο ε, αποσπάσαμε. Οπότε βεβαίω εντάξει, κάποια πράγματα θέλαμε να έχουν άλλο, αλλά νομίζω ότι γενικά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και εκφράζουμε την ικανοποίησή μα, την μεγάλη που έχουν τα πράγματα έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, ο πρόεδρο. Από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει κανεί το λόγο. Θέλετε να κλείσετε, κυρία Συγήτρια, πριν πούμε ποια είναι η προθεσμία για τι τροπολογίε. There is no deadline for amendments. Yeah, yeah, I know you're right. You're right. Just, just, just on the contrary. I was shocked. No, no, on the contrary. Just setting the. the... Όχι, Να πούμε τι γίνεται για, τις, ε, για, για, για την ψήφιση. Από ό,τι ξέρω, λες η ίδια, θα γίνει. Η ψηφορία δεν έχουμε ακούσει καμία αντίρρηση. Οπότε, δεν απομένει παρά να ευχαριστήσω την ε, γραμματεία μας και θα ψηφίσουμε στην Λίμπε στις 17 Θα Οπότε παρακαλώ να έρθετε όλοι. Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αλλά στις 3 ε, το απόγευμα, σε αυτήν την αίθουσα, θα κάνουμε την ε, ακρόασή μας, την έρευνα στις 3 το απόγευμα. Όμως έχουμε συνάντηση των συντονιστών αλλού. Σε άλλη αυτό για κάποιο λόγο. Στο 7C50. Στον 7ο όροφο αυτού του κτίριου. Όχι εδώ. Θα πάμε σε κάποια άλλη αυσό για τους συντονιστές. Στις 11.30 όπως έχουμε προγραμματίσει. Uh, really? The Αχ, συμπαθάτε μου, συμπαθάτε μου, λέει ο πρόεδρος. Από ό,τι μου είπαν, η συζήτηση για ε, την ακρόαση θα γίνει στο 6Q2, στο κτίριο Γιώζεφ Άνταλ. 6Q2. Εκεί πρόκειται να συζητήσουμε τα τη ε, έρευνας της Επιτροπής. Συγγνώμη για το ότι θα ξεβολευτούμε για να μετακομίσουμε εκεί. Ναι,